Ladies and gentlemen, good morning. It's Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Έχει περάσει η ώρα, ξεκινήσουμε λοιπόν τη συνάντησή μας. Το δεύτερο τμήμα της συνεδρίασης της Υποεπιτροπής ΣΕΝΤΕΡ. Προηγουμένως είχαμε την κοινή ανοιχτή δημόσια ακρόαση ε, με την ε, ομάδα Ντρουά για την χρήση των μη επανδρομένων αεροσκαφών και την καταπολέμηση της δημοκρατίας και τον ε, αντίκτυπο ω προ τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι κάτι το οποίο μα απασχόλησε κατά τη διάρκεια αυτή της ακρόαση. Τώρα θα περάσουμε στην τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής ΣΕΝΤΕΝ. Να σας υπενθυμίσω και πάλι ότι μεταδίδεται μέσω διαδικτύου η σημερινή συνεδρίαση. Ως προς ε, τη διερμηνία δίνεται προτίμηση στις ε, γλώσσες των πλήρων μελών της Υποπιτροπής Σέντε. Άμυνα και ασφάλεια. Θα ήθελα τώρα να υιοθετήσουμε την ημέρα διάταξη τη σημερινή συνεδρίαση. Αν συμφωνείτε κι εσεί, την εγκρίνουμε λοιπόν. Είναι πολύ μικρή η σημερινή ημέρα διάταξη. Μόλι ένα θέμα προ εξαιρετικά σημαντικό βέβαια. Εν ώψη και τη ε, διάσκεψη τη Βαρσοβία του ΝΑΤΟ που θα λάβει χώρα σύντομα. Στις 8 Ιουλίου θα ξεκινήσει. Ελήψη τυχών παρατηρήσεων. Θεωρώ ότι εγκρίνεται η μέση διάταξη. Ευχαριστώ. Να σας ζητήσω να εγκρίνουμε και τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης στις 30 Μαΐου. Εάν δεν υπάρχουν σχόλια, επιφυλάξεις μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, θα θεωρήσω ότι θα έχουν εγκριθεί και τα πρακτικά. Και τώρα επιτρέψτε μου να επηρεάσω στα σχόλια της Προέδρου και απευθείας λοιπόν να περάσουμε στο σημείο, το κύριο σημείο που θα μας προσχολήσει σήμερα, να καλωσορίσω θερμά τους διακεκριμένους ε, προσκεκλημένους μας. Ο κύριος Τζέμι είναι εδώ μαζί μας, ε, αναπληρωτής βοηθός Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ και περιμένουμε να ακούσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον ε, τα σχόλιά του και τις σκέψεις του για τη διάσκεψη της Βαρσοβίας. Και μετά θα έχουμε και ένα δεύτερο ομιλητή σήμερα. Το στρατηγό Ρόμαν Πόλκο. Ένα ιδιαίτερα πεπειραμένο στρατιωτικό, ιδίως ό,τι αφορά αποστολές σε πολλά μέρη του κόσμου όπου υπήρχαν ε, συμπλοκές και σειράξεις και Ο Πολωνό στρατηγό, πραγματικά συνέβαλε στην επίτευξη τη ειρήνη σε αυτέ τις περιοχές. Και εκπροσωπείται σήμερα και ένα πολύ γνωστό ίδρυμα, το γνωστό German Marshall Fund. Είναι εξαιρετικά πολύτιμη η συμβολή του ε, στις ε, διεργασίες μας. Σας ευχαριστώ και χωρίς επιπλέον καθυστέρηση να σας δώσω το λόγο αρχικά στον ε, γραμματέα Τζεμισία Σία για, για τα εισαγωγικά του σχόλια. Παρακαλώ, έχει το λόγο Τζέιμι. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε και εμένα, βεβαίω και τους δύο συναδέλφους μου εδώ σήμερα. Πάντα με μεγάλη μας χαρά ερχόμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χαίρομαι πολύ ότι υπάρχει και ένα κάποιο ενδιαφέρον εδώ στην αίθουσα για το ΝΑΤΟ που βεβαίω ε, δεν είναι και ασήμαντο εταίρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την προώθηση τη σταθερότητα στην Ήπειρο μα και εν γέννη την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια. Σα ευχαριστώ λοιπόν για την παρουσία σα και το ενδιαφέρον σα. Ξέρω ότι πρέπει να είμαστε σύντομοι στα εισαγωγικά μα ε, σχόλια, αλλά θα δυσκολευτώ λίγο. Γιατί οι διασκέψει του ΝΑΤΟ δεν λαμβάνουν χώρα τόσο συχνά όσο ε, οι ευρωπαϊκές σύνοδοι κορυφής. Ε, δεν είναι πολιτική κριτική αυτό. Έτσι είναι τα πράγματα. Κάθε δύο χρόνια συναντιόμαστε και αυτό γιατί ε, Είχαμε και πριν από δύο χρόνια στην Ουαλία, το Σεπτέμβριο του 2014, την τελευταία τέτοια σύνοδο κορυφή και από τότε έχουμε πολλέ νέε εξελίξει, πολλέ νέε πρωτοβουλίε και αντί να ασχοληθούμε με ένα-δύο ζητήματα η Σύνοδος Κορυφής θα πρέπει να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα ζητήματα. Πολλά μέτωπα δηλαδή, από την Ανατολή και την επανανάντηση της ε, Ρωσίας, αλλά και για τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και όλες τις αλλαγές ε, που έχουν επέλθει. Θα δείτε λοιπόν ότι έχουμε ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων ε, που θα μας απασχολήσουν και θα πρέπει να εξετάσουμε. Σε ένα βαθμό λοιπόν είμαστε υποχρεωμένοι, χωρίς να μείνουμε εδώ βεβαίως μέχρι το βράδυ, κάπως θα πρέπει να τα διατρέξω όλα αυτά πολύ σύντομα και επιγραμματικά. Και ελπίζω, κυρία Πρόεδρε, στη συνέχεια να περάσουμε σε, μια, σε βάθος ανάλυση αυτών των ζητημάτων που σας ενδιαφέρουν ιδιαίτερως. Επομένως, κάντε λίγη υπομονή, καθώς θα διατρέχω όλη την ημέρα στη διάταξη της Συνόδου Κορυφής. Για να σας βοηθήσω όμως, Υπάρχουν ε, δύο μεγάλες θεματικές ε, ενότητες. Το ένα είναι η άμυνα και η αποτροπή σε ό,τι αφορά την επαναγκαθίδρυση ενός ε, κατάλληλου συστήματος ασφάλειας και αποτροπής στο ΝΑΤΟ για να διατηρήσουμε την ειρήνη που έχουμε εδώ και 50 χρόνια περίπου σε ό,τι αφορά την ακαιρεότητα τουλάχιστον των μελών του ΝΑΤΟ. Το δεύτερο είναι σε ό,τι αφορά τη σταθερότητα, την προαγωγή της σταθερότητας που αφορά άλλες πτυχές και τις χώρες του ΝΑΤΟ αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας ασχοληθούμε λοιπόν πρώτα με την άμυνα και αποτροπή. Λόγω και της ε, τοποθεσίας που θα λάβει χώρες με τους κορυφείς, η Βαρσοβία δηλαδή, θα είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει ιδιαίτερως. Εδώ έχουμε δύο κύρια στοιχεία. Πρώτον, η υλοποίηση των αποφάσεων που ελήφθησαν στην Ουαλία. Ε, απαιτείται και μια αξιοπιστία εδώ πέρα, ότι τα τελευταία δύο χρόνια κάναμε αυτά που μας ζητήσατε να κάνουμε στην περασμένη συνάντηση. Κάναμε δηλαδή σωστά τη δουλειά μας. Και εδώ από την Ουαλία προέκυψε ένα σχέδιο δράσης ετοιμότητας για να καλύψουμε το κενό, τουλάχιστον ό,τι αφορά τη, τις δυνατότητες, την ικανότητα του ΝΑΤΟ ε, στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη σε μια εποχή ε, που ε, η Ρωσία προσήρτησε την Κρυμαία και ανέπτυξε τις δυνάμεις της για να αποσταθεροποιήσει την Ανατολική Ουκρανία. Τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού του σχεδίου δράσης ετοιμότητας έχουν υλοποιηθεί. Είχαμε μία κοινή task force πολύ υψηλής ετοιμότητας με επιμέρους ε, δυνάμεις ε, τα έχουμε πιστοποιήσει είναι έτοιμη αυτή η ταξιαρχία ε, να αναπτυχθεί. Έχουμε διπλασιάσει το μέγεθος της task force αυτής από το μέγεθος της ταξιαρχίας και περάσει το μέγεθος της δημιουργίας θα δούμε όμως ποια θα είναι κατάλληλη μορφή με περισσότερα θαλάσσια, εναέρια ή χερσαία μέσα. Αυτό δεν αφορά μόνο την ανατολική πλευρά, ε, μπορεί να υλοποιηθεί ενδεχομένως και στο νότο. Έχουμε πιο πολλά ε, διεθνή αρχηγία στα κράτη-μέλη μας στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη. Θέλουμε να έχουμε υποδομές υποδοχής για τις νεοφυκτήσεις ε, δυνάμεις. Έχουμε αναβαθμίσει τη στήριξή μας στην Πολωνία, στη Δανία και έχουμε πλέον ε, διεθνή αρχηγία για ε, τα βορειοανατολικά. Και βλέπετε, γιατί φαντάζομαι όλοι τα έχετε διαβάσει ε, στις εφημερίδες, στην τηλεόραση, ότι έχουμε αναπτύξει τις δυνατότητες ασκήσεων και ανάπτυξης. Είχαμε 300 τέτοιες σχετικές πρωτοβουλίες και ασκήσεις πέρυσι η πιο σημαντική ήταν η, η, transjuncture. Εντάξει, τώρα αυτός είναι στρατικός ε, όρος που έλαβε χώρα στην Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ιταλία πέρυσι το φθινόπωρο. Η μεγαλύτερη κοινή άσκηση του ΝΑΤΟ εδώ και δεκαετίες, με 36.000 στρατιώτες. Όμως αυτό ήταν για να καταδείξουμε ότι αν είναι απαραίτητο, μπορούμε να επανέλθουμε σε αυτές τις μεγάλες κλίμακας επιχειρήσεις. Όλα αυτά βεβαίως ε, για να αποστείλουμε το μήνυμα της ε, αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ ότι ε, παίρνουμε πολύ στα σοβαρά την δέσμευσή μας που προκύπτει από το άρθρο 5 για την υπεράσπιση των κρατών μελών μας. Όμω δεν θέλουμε να προκαλέσουμε και να κλιμακώσουμε την ένταση. Έχουμε καλέσει τους Ρώσου σε όλες τις ασκήσει μα. Μακάρι να έκαναν και εκείνοι το ίδιο και να μας προσκαλούσαν να παρευρεθούμε στις δικές τους έχουμε διατηρήσει την πολιτική δέσμευση που κάναμε το 1997 στη Ρωσία να μην θέσουμε ε, ε, πυρηνικά όπλα, πολύ σημαντικές θεωρητικές δυνάμεις στα, ε, στην επικράτεια των νέων κρατών μελών. Πάντα στο ΝΑΤΟ κάνουμε το ελάχιστο που θεωρούμε ότι απαιτείται για να διατηρήσουμε την αξιοπιστία της κοινή μας υπεράσπισης και άμυνας. Η δεύτερη σημαντική πτυχή της υλοποίησης των αποτελεσμάτων της Συνόδου Κορυφής της Ουαλίας είναι το πώς θα ε, σταματήσουμε κάπως τις συνεχούμενες περικοπές ε, στις δαπάνες αμήνης. Στο 2% είχαμε ε, ορίσει το όριο σε ό,τι αφορά την άμυνα και 20% του προϋπολογισμού της άμυνας για τον εξαφανισμό. Προφανώ δεν περιμένετε να πω ότι όλοι οι εταίροι έχουν επιτύχει αυτόν τον ε, στόχο, γιατί βεβαίω και η οικονομική κατάσταση, ιδίω εδώ στην Ευρώπη, ήταν πολύ πιεστική και αρνητική. Το γνωρίζουμε και πράγματι μετά την Ιουαλία, από τους τέσσερις ε, συμμάχους που δαπανούσαν το 2% του ε, ΑΕΠ στην άμυνα, έχουμε περάσει στους πέντε συμμάχους η Πολωνία, για παράδειγμα, είναι η πέμπτη αυτή χώρα με πολύ σημαντικέ προσπάθειε. Είναι ενθαρρυντικά μα τα στοιχεία. Πλέον έχουμε 17 συμμάχου. Η μεγάλη πλειοψηφία που έχουν αυξήσει του αμυντικού του προπολογισμού από το 2014 και μετά. Σήμερα έχουμε 12 ε, συμμάχου που μα έχουν δώσει ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό για να περάσουν μέσα στην επόμενη δεκαετία στο 2% του ΑΕΠ. Χώρε όπω η Γαλλία έχουν σταματήσει τι περικοπέ στον αμυντικό προπολογισμό και έχουν επανέλθει σε προηγούμενα επίπεδα δαπανών. Έχουμε δύο επιπλέον συμμάχου, από του 7 στου 9, έχουμε περάσει στο 20, που έχουν περάσει σε αυτό το 20%. Θα ήθελε ο Γενικό Γραμματέα Τόντομπερκ κάτι παραπάνω, βεβαίω και γι' αυτό και θα συνεχίσει να το επιδιώκει. Αλλά τουλάχιστον σταματούμε αυτή την ε, πτώση, τη φθήνουσα πορεία. Και αυτό είναι θετικό, γιατί είναι εθνικέ αυτέ οι δυνάμει. Βεβαίω ε, συμμετέχουν στο ΝΑΤΟ, όλο αυτό το επιπλέον στρατιωτικό δυναμικό, η ικανότητα που δημιουργείται, ε, οδηγεί και σε καλύτερη ετοιμότητα, ενδεχομένως και καλύτερη ικανότητα για το CSDP, για την ΠΑΚ, Κοινή Πολιτική Ασφάλειας. Ε, δεν ξέρουμε κατά πόσο η έκθεση θα είναι αρνητική για την ΟΛΕΑ. δεν νομίζουμε ότι θα είναι αυτό, αλλά μετά την Ουαλία, η στάση της Ρωσίας ως προς τη συμμαχία και η δυναμική που έχει διαμορφώσει με αυτές τις ε, απρόβλεπτες ασκήσεις, για παράδειγμα, προκλητικές ε, κινήσεις με τα, ε, απέναντι στα ανατοϊκά σκάφη, για παράδειγμα, σημαίνει ότι πρέπει να δώσουμε πλέον διασφαλίσεις στους ε, συμμάχους μας από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Πρέπει με, με μια ήπια αλλά σημαντική ε, τροποποίηση να επαναφέρουμε την ισορροπία που υπάρχει ε, Επομένω, ε, ο βασικό τίτλο, αν θέλετε, τη εφημερίδα την επόμενη εβδομάδα στην Ουαλία θα είναι ε, η θέσπιση αυτών των τεσσάρων πολυεθνικών ταξιαρχιών από την Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και θα ανακοινωθεί και το τέταρτο τέτοιο κράτος που θα αναλάβει αυτή την ηγετική θέση. Θέλουμε όμως εκ περιτροπή ε, να κινούνται αυτές οι μονάδες και αυτό γιατί θα έχουμε τη μέγιστη δυνατή κατάρτιση για τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό ε, στρατιωτικών δυνάμεων με τη μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία. Αλλά ανα πάσα στιγμή ε, το ίμιση των ατοικών δυνάμεων θα αναπτύσσεται και αυτό θα δίνει το σημάδι, το μήνυμα ότι το να επιτεθεί κανείς σε έναν ισούται με την επίθεση σε όλους ουσιαστικά. Εντάξει, τώρα είναι πολλές λεπτομέρειες, δεν θέλω να σας κουράσω, όμως θα εξετάσουμε ε, την ε, δομή μας. Ε, αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε πολλές μονάδες που θα πρέπει να συντονίσουμε, τα προγράμματά μας, την διασύνδεση μεταξύ των τοπικών δυνάμεων, γιατί και στην Πολωνία υπάρχει σημαντική δύναμη να υπάρχουν περισσότερες τοπικές δυνάμεις και αναπληρωματικές. εξετάσουμε το θέμα A2AD και την ε, πρόσβαση, τη δυνατότητα πρόσβαση σε, όλη μας την επικράτεια, ανα πάσα στιγμή, χωρίς προσκόμματα, χωρίς ε, επιπλοκές. Και βεβαίω θα πρέπει να εξετάσουμε και τη διάρθρωση μεταξύ των επιτόπιων δυνάμεων και το πόσο γρήγορα ε, και αποτελεσματικά μπορούμε να αναπτύξουμε τις ε, δυνάμει μα. ούτω ώστε να μην υπάρξουν κενά στην δομή την οποία θα αναπτύσσουμε. Όλα αυτά όμως μόνο για αποτρεπτικούς σκοπούς. Θέλουμε λοιπόν να κάνουμε τις προσπάθειες για να δείξουμε την, ε, τις δυνατότητες ε, αποτρεπτικές. Όμως θέλουμε να καταδείξουμε και την ύφεση εδώ. Πώς δηλαδή θα οδηγηθούμε προς έναν πιο ε, παραγωγικό και επικαδηματικό διάλογο με τη Ρωσία. Όταν η Ρωσία βεβαίω δει και πιστεί ότι το ΝΑΤΟ δεν πρόκειται να αφήσει να εκφοβίζεται από τη Ρωσία και ότι είναι, πρόκειται για ένα αμοιβαίο συμφέρον ε, τη διαφάνεια, ε, τη σταθερότητα και των μια κοινή προσπάθεια και από του δύο. Πρέπει λοιπόν πέραν τη αποτροπή να εξετάσουμε και την ύφεση. Κάτι άλλο το οποίο μας απασχολεί είναι οι υβριδικές μορφές πολέμου. Είτε μας αρέσει ο όρος είτε όχι, ξέρετε τι εννοούμε. Μη συμβατικές, μη γραμμικές ε, τακτικές και μέθοδοι. Ε, κυβερνοεπιθέσεις, στρατηγικές επιχειρήσεις ε, άμυνας και επικοινωνιών. Πρέπει να είμαστε πραγματικά σε εγρήγορση σε ό,τι αφορά την αποσταθεροποίηση όσο θα ήμασταν και με μια κανονική στρατιωτική επίθεση. Και εδώ θεωρούμε ότι είναι κρίσιμη σημασία η Ευρωπαϊκή Ένωση και όπω ξέρουμε, ε, μαζί με τον Γενικό Γραμματεία και την ε, κυρία Φεντερίκα Μογκερίνη, ε, σχεδιάζουμε μια κοινή διακήρυξη στη Βαρσοβία για τη συνεργασία ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλά έχουν γίνει και σε επίπεδο επιτελείων σε ό,τι αφορά τι επαφέ στον κυβερνοχώρο συμφωνία μεταξύ των επιμέρου υπηρεσιών μα, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, εγχειρίδια. Αυτό σημαίνει ότι με στενισμένο δρόμο εξετάζουμε και από τι δύο πλευρέ ε, το πώ θα ακριβώ θα χειριστούμε την ανάπτυξη των υβριδικών μορφών πολέμου σε διάφορα σενάρια και ποια, ο ποιο οργανισμό είναι σε καλύτερη θέση να αντιμετωπίσει το κάθε γεγονό και περίσταση. Επίγνωση τη κατάσταση και χρειαζόμαστε και ασκήσει, καθώ ε, θα απομακρυνόμαστε μετά από τη Βαρσοβία, Σκοπός μας θα ήταν να προσχωρήσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση κατευθείαν στην Βαρσοβία, αλλά τουλάχιστον υπάρχουν κοινέ συντονισμένε εσκήσεις και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τον ΝΑΤΟ. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τώρα σε περίοδου ε, Ειρηνή. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση να σας προσθέσω ότι δεν θέλουμε συνεργασία ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης να περιοριστεί στον υβριδικό πόλεμο, παρότι αναγνωρίζουμε το κοινό ενδιαφέρον. Το ΝΑΤΟ τους τελευταίους μήνες έχει υπογράψει μία ε, συμφωνία με τη Frontex, την πρώτη στην ιστορία μα, ούτω ώστε να επιμεριζόμαστε πληροφορίε για το Αιγαίο, καθώς έχουμε αναπτύξει μία ναυτική δύναμη στο Αιγαίο και συντονισμό ανάμεσα στην ε, Ελλάδα και στην Τουρκία. Είναι μια μεγάλη επιτυχία αυτή και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία στην Κεντρική Μεσόγειο ε, μετά τη Λιβύη, μετά την κρίση τη μεταναστευτική και το προσφυγικό. Ε, υποστηρίζουμε τη, Σοφία, και ό,τι κάνει στην, στην Μεσόγειο ε, για να περιοριστεί η ροή των μεταναστών και για πιο ανθρωπιστικές επιχειρήσεις. <clears throat> Στη Σόφια ε, σώσαμε μερικούς ανθρώπους που θα μπορούσαν να είχαν να πνιγεί Είναι πολύ σημαντικό Ε, να περάσουμε ε, σε μεγαλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών. Έχουμε δορυφόρους, έχουμε ανεπάνδρωτα ελικόπτερα. Έχουμε ε, επίσης τα ελικόπτερα πάρα πολύ προχωρημένης τεχνολογίας με κοινό στρατιωτικό δυναμικό. Έχουμε ε, τον ΕΚ, το Αμερικανικό Στόλο, ε, την κοινή διοίκηση, έχουμε αεροσκάφη, μαχητικά αεροσκάφη κτλ. Και θα θέλαμε με το διάλογο αυτό με την Ευρωπαϊκή Ένωση να συγκεντρώσουμε αυτές τις, ε, αυτό το δυναμικό, το δικό μας και το δικό σας. Όπως κάναμε με την αντιμετώπιση της πειρατείας πριν από μερικά χρόνια. Τώρα, να περάσω σε ένα άλλο μεγάλο θέμα. Ε, ο Νότος είναι διαφορετικός βέβαια από την Ανατολή. Ε, τα θέματα δεν είναι, αυτά δεν είναι γραμμικά, δεν μπορεί να δώσει γραμμική απάντηση. Κάθε χώρα είναι διαφορετική ε, και έχουμε πολλές διαφορετικές προκλήσεις που αλληλεπιδρούν με αρνητικό τρόπο. Ε, πρέπει να αναγνωρίσουμε το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να είναι ο μόνος φορέα ή ο πρωταρχικό φορέα. Φυσικά έχουμε υψηλό προφίλ. Ε, στην, Ανατολή, στην ανατολική πλευρά μας έχουμε την κλασική αποτρεπτική δύναμη. αλλά στους, έχουμε τους νότιους συμμάχους που είναι και μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Ε, το ISIL ε, πειραματίζεται με χημικά όπλα. Ε, υπάρχουν, ας πούμε, χαμηλής έντασης απειλές. Ε, στο μέλλον μπορεί να αποκτήσει κρατικού τύπου, ας πούμε, ε, ισχύ. Θα πρέπει να γνωρίζουμε όλες αυτές τις απειλές και φυσικά η αρχική ενεργοποίηση ε, του την επόμενη εβδομάδα στη Βαρσοβία ε, του πυραυλικού αμυντικού ε, δυναμικού ε, θα καλύψει όλους τους νότιους εταίρους μας και την Τουρκία εναντίον των πυραυλικών απειλών. Επίσης θα πρέπει να βοηθήσουμε τη συμμαχία κατά του ISIS όπου μπορούμε να επεκτείνουμε τα αεροσκάφη AWACS ούτως ώστε να υπάρξει μια συνειδητοποίηση του κινδύνου και θέλουμε επίσης να αυξήσουμε περισσότερο το αμυντικό δυναμικό στο Νότο. Ε, έχουμε ήδη project ε, ε, με, το Ιράκ, με την Ιορδανία. θέλουμε επίσης να επιστρέψουμε στη Βαγδάτη και να δώσουμε κατάρτιση και μαθήματα κτλ. Ε, ε, τελευταίο σχόλιο για την, στα πλαίσια της ΚΠΑ. Υπάρχει μεγάλη πραγματογνωμοσύνη. Ε, κοιτάξτε την ε, Λιβύη, όπου προφανώ ε, έχουμε συμφέρον να συνεργαστούμε. Θα θέλαμε μια συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να δούμε πώ μπορούμε να συνενώσουμε με συμπληρωματικό τρόπο το, το αμυντικό μα δυναμικό, ε, ούτω ώστε να μην ξοδεύουμε χρήματα σε μαύρε τρύπε, συγκεντρώνοντα τι προσπάθειέ μα εκεί που έχει νόημα για, για τι τοπικέ δυνάμει, ε, εκεί όπου οι τοπικέ δυνάμει είναι βιώσιμε. Γιατί μόλις ε, φεύγεις, ας πούμε, μερικές φορές ε, όλα τα δισεκατομμύρια που, που έχεις δώσει ε, είναι σαν να μην τα έχεις δώσει ποτέ, ας πούμε. Θα πρέπει να υπάρχει μια βιωσιμότητα, μια συνέχεια. αυτή είναι η γεύση, ας πούμε, που θα ήθελα να σας δώσω. Δεν τα ανέφερα όλα το λέω προς ανακούφισή σας. Πάντως σας το λέω για να σας πω ότι αυτό δεν είναι κλασική, ε, κλασικός τρόπος ε, λειτουργίας. Είναι ιστορική ε, σύνοδος ε, του ΝΑΤΟ και σε μια χρονική στιγμή όπου ε, τα νέα είναι αρκετά δυσίωνα τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες και η συνοχή της Ευρώπης και της Διατλαντικής Συμμαχίας αμφισβητείται. Σωστό ή λάθος από πολλούς. Και το σημαντικό που θα προκύψει ε, από τη Βαρσοβία, πέρα από τα συγκεκριμένα που θα κάνουμε, είναι αυτή η αίσθηση ενότητας, σκοπού και αποτελεσματικότητας ε, από πλευράς ε, της διατλαντική κοινότητα. Ότι μπορούμε δηλαδή να ελέγξουμε την κατάσταση, ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα. Είναι δύσκολη κατάσταση, δύσκολη συγκυρία, αλλά δεν πρόκειται να διαιρεθούμε. Και δεν σας λέω ότι η Βαρσοβία από μόνη της θα δημιουργήσει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην Ήπειρο, κάτι που χρειαζόμαστε αλλά μετά από τόσα ε, κακά νέα, το ένα μετά το άλλο, καλό θα ήταν να ακούσουμε και κάτι καλό για μια φορά. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου δώσατε τη δυνατότητα να έρθω εδώ και να μιλήσω στο Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστούμε, κύριε Γραμματέα Πραγματικά ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η παρέμβασή σας και πάρα πολύ ενθαρρυντική. Σας ευχαριστώ. Και τώρα θα ήθελα να ζητήσω από τον στρατηγό και να πάρει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ και καλημέρα σας. Ο Ρόμαν Πολκο ονομάζομαι και θα ήθελα να σας αναφέρω και να κάνω κάποια σχόλια για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Πρώτο περάσω όμως ε, στα σχόλια μου αυτά θα ήθελα να σας αναφέρω ότι πρόκειται για το 18ο έτος συμμετοχής μας στο ΝΑΤΟ. Πριν από 18 χρόνια, λοιπόν, ήμουν διοικητής μιας ε, ε, δύναμης εγκυρής απόκρισης, η οποία ιδρύθηκε και τότε. Ήμασταν ιδιαίτερα ε, έτοιμοι να μετακινηθούμε και το σύμβολό μας ήταν η γροθιά. Χαίρομαι ιδιαίτερα λοιπόν που σήμερα μπορώ να σας μιλήσω για το τι προτίθεται να κάνει το ΝΑΤΟ και θα συζητήσουμε λοιπόν διάφορους τομείς κατά την διάρκεια της Συνόδου. σταθεροποίηση εκτός της επικρατείας μας και ενσωμάτωση, ενοποίηση του ΝΑΤΟ και ενοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρώτος τομέας. Εδώ έχουμε να φέρουμε πολλά θετικά στοιχεία. Διοργανώθηκαν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες επιχειρήσεις, περιλαμβάνοντας πάνω από 30.000 στρατιώτες. Οι ασκήσεις λοιπόν αυτές ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες, γιατί το σενάριο δεν ήταν προκαθορισμένο. Και μου θύμισε τον ε, Βρετανό στρατηγό Ράιτ. Η κατάσταση λοιπόν η οποία διαμορφώθηκε ήταν η εξή. Ήμασταν αντιμέτωποι ε, ε, έξαφνα με ένα αναπάντεχο σενάριο. Αυτή ήταν η προσωμείωση, όπως και αναμένουμε σήμερα από την ε, Ρωσία. Και έτσι προσωμιώσαμε λοιπόν ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις ε, στον άμαχο πληθυσμό, στα γυναικόπαιδα και έτσι λοιπόν ε, ήταν πάρα πολύ ωφέλιμη αυτή η προετοιμασία. Εξακολουθούν ασφαλώς να υπάρχουν ακόμα κενά και προβλήματα. Αλλά, όπως λέμε και στη στρατιωτική ορολογία, από τη στιγμή που εντοπίζεται ένα κενό, ουσιαστικά δεν υπάρχει πλέον. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να υπάρχει ομοιογένεια, να υπάρχει ένα ενιαίος χαρακτήρας. Μετά λοιπόν την σύντομη διεξαγωγή των ασκήσεων αυτών ε, έγιναν και δηλώσει από κάποιου εταίρου. Ακούσαμε ότι πρόκειται για μια περιττή πρόκληση, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν βοηθά σε περίπτωση συγκριουσιών. Το άρθρο 3, ωστόσο, της συνθήκης του ΝΑΤΟ αναφέρει ότι η ανάπτυξη των μεμονωμένων και συνολικών συλλογικών ε, δυνατοτήτων και ικανοτήτων άμυνας είναι απαραίτητο, γιατί αυτό συναποτελεί τη συνολική αμυντική ικανότητα. Τέτοιες ασκήσεις, λοιπόν, θα πρέπει να γίνουν ρουτίνα, δεν αποτελούν πρόκληση. Τέτοιες λοιπόν οι ικανότητες άμυνας σε καμία περίπτωση δεν θα μπορέσουν να αναπτυχθούν και τώρα, στο σκέλος της επικοινωνίας, η επικοινωνία τονίζω, γιατί δεν αρκεί η ενημέρωση. Η ενημέρωση από μόνη της είναι άχρηστη, αν δεν διαβιβάζεται η πληροφορία. Και αν θέλουμε πραγματικά να έχουμε σωστές ικανότητες αποτροπής θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει τη σωστή επικοινωνία. Μια δεύτερη σημαντική πρόκληση έγινε στο εξή ε, τομέα. Καταπολέμηση του Ισλαμικού κράτους, καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ε, οι Ρώσοι στρατιώτε, ε, οι άνθρωποι με τα πράσινα όπως αναφέρονται. Παρατηρήσαμε λοιπόν στο... και στη Μέση Ανατολή και στο Ιράκ ότι προέρχονται πάρα πολλά προβλήματα και μετά από την απόσυρσή τους. Και ότι είναι πάρα πολύ σημαντική ασφαλώς η ανάπτυξη των ενδογενών δυνάμεων και ότι χρειάζεται και μια αλφα στοχοθέτηση διαρκώς. Χρειάζεται ένα σενάριο, ένα όρεμα για την περίοδο μετά την αποχώρηση των δυνάμεων. Μία αποστολή σκέτη χωρίς ένα σενάριο για το μετά ε, αποτελεί ένα φιάλτη, όπως είπε και ένας ε, Αμερικανός αξιωματικός. Άρα, σε ό,τι αφορά τις μελλοντικέ προκλήσεις, είναι σημαντικό να σκεφτούμε σε βάθος χρόνου πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Γιατί αν δεν υπάρχει μια κοινή στρατηγική, αν δεν έχει καταρτιστεί μια κοινή στρατηγική, μπορεί να δοθεί μάλιστα και η εντύπωση ότι κάθε ε, δυτικό κράτο ε, έχει και τον αγαπημένο του δικτάτορα στην περιοχή, τον οποίο και υποστηρίζει. Ο Άσάντα αποτελεί ένα καλό παράδειγμα. Γιατί πολλές ε, χώρες θεωρούν ότι πρόκειται για μια προσωπικότητα η οποία πρόκειται να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Αναρωτιόμαστε λοιπόν ποιο είναι πιο επικίνδυνο, ο Ασάντ ή το Ισλαμικό κράτο και τελικά ποιο οφείλεται για το μεγάλο κύμα των προσφύγων. Τώρα, σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση τη τρομοκρατία, στο σημείο αυτό θα πρέπει να υπάρχει μια ενιαία επικοινωνία από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Χρειάζεται μια κοινή στρατηγική. Και θα πρέπει να δράσουμε από κοινού. Μόνο τότε θα μπορέσουμε να έχουμε κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα. Δεν είναι δυνατόν κάθε κράτο να ακολουθεί τα εθνικά του συμφέροντα. Γιατί πολύ απλά στην περίπτωση αυτή δεν θα είμαστε σε θέση ως συμμαχία να δράσουμε. Ένα τρίτο σημαντικό θέμα, η ενοποίηση του ίδιου του ΝΑΤΟ. Η ενοποίηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεδομένων και των προσφάτων ε, δεδομένων και περιστατικών, ιδιαίτερω και του Brexit, αναρωτιέμαι κατά πόσον μπορεί να υπάρξει το ΝΑΤΟ χωρί την αγγλική γλώσσα. Δεν μπορώ να φανταστώ το ΝΑΤΟ χωρίς αγγλικά. Δεν ξορίζω και κάποια άλλη ε, στρατιωτική γλώσσα πέρα από τα αγγλικά. Ακόμα και στην πολυνική γλώσσα χρησιμοποιούμε αγγλικά ακρονίμια, αγγλική ορολογία. Αυτή η ορολογία λοιπόν δύσκολα μπορεί να μεταφραστεί και να μεταφερθεί σε άλλη γλώσσα. Η ε, ΙΠΑ εδώ και καιρό ζητούν να αναλάβει τις ευθύνες της η Ευρώπη και να αναπτυχθούν ε, δυνάμεις και ικανότητες άμυνας. Γιατί το δεύτερο σκέλος της ΚΕΠΑ αναφέρεται στην άμυνα. Στην Πολωνία, λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι έχουμε αναπτύξει τέτοιο δυναμικό και θέλουμε να ξεπεράσουμε και τα προδιαγραμμένα επίπεδα. Τι γίνεται, λοιπόν, σε ό,τι αφορά τη συνολική Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ικανότητες άμυνα. Υπάρχουν αξιώσει για τέτοιες δυνάμεις. Το θέμα, λοιπόν, όμως, είναι πώς θα δημορφωθούν οι δυνάμεις αυτές, πώς θα χρηματοδοτηθούν, ε, ποιος θα τις προστάζει και πώς θα ε, έχουν, ε, τι σχέσεις θα έχουν με τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ. Θα υπάρχουν συνέργειες, συμπληρωματικότητα, θα προκληθούν τριβές, το οποίο ασφαλώς θα έχει και αρνητικές επιπτώσεις στις αμυντικές μας ικανότητες. Στο ίδιο το ΝΑΤΟ τώρα λοιπόν, το μεγάλο ερώτημα είναι η αποφασιστικότητα. Οι αποστολή στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ κατέδειξαν με σαφήνεια πού βρίσκονται τα όρια μας. διατίθεται δυνάμεις, αλλά πάντα υπάρχει ένα ανώτατο όριο. Είναι δύσκολο λοιπόν να υπάρξει μια κεντρική διοίκηση των στρατευμάτων αυτών με περιορισμένες ικανότητες και με εθνικά, με εθνικούς περιορισμούς. Μια δεύτερη μεγάλη πρόκληση για όλους τους συμμάχους είναι το τι αποτελεί επίθεση. Ποια επίθεση θέλετε ευρετική επίθεση και από ποιο σημείο και πέρα μπορούμε πραγματικά να πούμε ότι χρειάζεται μια συνολική πλήρους ανάπτυξης αντίδραση γιατί πρόκειται για πόλεμο. Έχουμε πόλεμο ενημέρωσης, ενέργειας, προπαγάνδας. Όλα αυτά υφίστανται. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι ο πόλεμος σήμερα έχει πάρα πολλές μορφές και έχει καταστεί τόσο περίπλοκος που πρέπει να ειδωθεί Συνολικά, συνοψίζοντα, πρέπει να σα πω ότι αντιμετωπίζουμε πάρα πολλέ προκλήσει και πάρα πολλού κινδύνου. Καταρχά, έχουμε έναν ε, Πούτιν ο οποίο δεν μπορεί να προβλεφθεί πώ θα αντιδράσει. Πολλοί τον θεωρούν πρόβλημα, αλλά και πολλοί τον θεωρούν και λύση του προβλήματο. Έχουμε το Ισλαμικό κράτο, αποτελεί μια μεγάλη, ένα μεγάλο ρίσκο, ένα μεγάλο κίνδυνο και εδώ χρειάζονται στρατηγικέ. Η στρατηγική του 2010 είναι παροχημένη πλέον. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια νέα βάση για την ανάπτυξη των δράσεών μα και των ενεργειών μα και θα πρέπει αναλυτικά να προσεγγίσουμε το θέμα αυτό. Δεν είναι δυνατόν να αφήνουμε το θέμα αυτό σε γραφειοκράτε οι οποίε ε, θέλουν απλά να ολοκληρωθεί έτσι η σύνοδο Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, λέει πρόεδρο. Σα Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να είμαι εδώ σήμερα μαζί σας με τους συγκεκριμένους ε, συναδέλφους μου. Πολλά έχουν ήδη υποθεί, επομένω δεν θέλω ε, να επαναλάβω τα ίδια και τα ίδια Όμως, όπως θα καταλάβετε μάλλον, είμαι Αμερικανό ε, πολίτης. Το German Marshall Fund είναι German Marshall Fund των Ηνωμένων Πολιτειών. Είμαστε Αμερικανοί λοιπόν, παρότι έχουμε αυτή την ιστορική σύνδεση στην Ευρώπη. Τώρα θα ήθελα να πω δύο λόγια, ε, συνεχίζοντας κατά κάποιον τρόπο από εκεί που σταμάτησε ο Τζέμι Σέι. Ε, ζητήματα που άπτονται της ε, γενικότερης εικόνας που εξετάζουμε και άλλα που θα είναι ανοιχτά, εκκρεμή ζητήματα στη συνέχεια. Τρεις είναι οι βασικές μου παρατηρήσεις. Το πρώτο αφορά τα επίπεδα φιλοδοξίας της Συνόδου Κορυφής. Πόσο φιλόδοξη και πόσο σημαντική θα είναι τελικά υπήρχε ένας φόβος ότι ε, δεν θα κάνουμε αρκετά όσα δηλαδή απαιτούν οι περιστάσεις. Και Τζέμι τελικά προκύπτει ότι θα κάνει πολλά. Ε, δεν έχει σκοπό να διαμορφώσει μια νέα στρατηγική έννοια και πλαίσιο. Αυτό θα γίνει στην πορεία. Όμω ε, είναι πολλά τα στοιχεία στη μεσαδιάταξη. Κανεί νομίζω δεν θα μείνει απαγοητευμένο. Είναι αρκετά φιλόδοξη λοιπόν η Σύνοδο Κορυφή. Κατά τη γνώμη μου, είναι μεγάλο πειρασμό να εξετάσουμε την στρατηγική του ΝΑΤΟ ω μία σειρά διαχείριση κρίσεων. Είναι αυτό, αλλά είναι κάτι πολύ παραπάνω. Η πρόκληση τη προσαρμογή είναι αυτή για τον ΝΑΤΟ, αλλά και ω προ ε, την παγκόσμια στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση που μόλις δημοσιοποιήθηκε, υπερβαίνουν κατά πολύ αυτό ακριβώς το στοιχείο. Αν δείτε τα όσα έχουν ήδη περιγράψει συνάδελφοι στην Ανατολή ή στον Νότο, δεν μιλούμε μόνο για ζητήματα διαχείρισης κρίσεων, θα εξετάσουμε και θα αντιμετωπίζουμε αυτές τις κρίσεις για πολλά χρόνια ακόμα και ενδέχεται να μην, να μην επιληθούν για πολλά χρόνια ακόμα. Αυτό είναι ένα νέο στοιχείο λοιπόν. Δεν νομίζω ότι η ένταση ε, με την Ρωσία και η επιδείνωση των σχέσεων με τη Ρωσία θα φύγει, θα εξαφανιστεί σύντομα, ενδεχομένως να μετριαστεί αλλά δεν θα επανέλθουν οι σχέσει σύντομα. Και πλέον η Ρωσία έχει και έναν πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει. Προ τον Νότο τώρα και πάλι δεν βλέπω πραγματικέ προοπτικέ ε, επίλυση ζητημάτων. Ουσιαστικά μπορούμε να έχουμε και δεκαετίες χάου και ανοιχτή ε, σύραξης. Αυτή είναι μια τεράστια πρόκληση και έχει μια απλή διαχείριση κρίσεων. Και έτσι, ουσιαστικά και το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση το εξετάζουν ως ένα στρατηγικό πρόβλημα. Το δεύτερο που ήθελα να πω είναι κάτι το οποίο έχει ήδη αναφερθεί. Πώς το ΝΑΤΟ εξισορροπεί Ανατολή, Νότο, ίσως και τον Βορρά. Εντάξει, μπορεί να μην μιλήσουμε για την Αρκτική, αλλά είναι σημαντικό ζήτημα, ιδίω ε, για χώρε όπως η Νορβηγία. Ε, Πώ γίνεται αυτή η ισορρόπηση μεταξύ Ανατολή και Νότου, λοιπόν. Αναπόφευκτα θα επικεντρωθούμε κυρίω στη Σύνοδο Κορυφή στην Ανατολή. Αυτό ενδεχομένω γιατί είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Όπω ανέφερε και ο στρατηγό. Όμω θεωρώ ότι τα εκρεμή ζητήματα από τη Σύνοδο Κορυφή μάλλον θα αφορούν τον Νότο. Και θα μα πάρει χρόνο να τα επιλύσουμε όλα αυτά. Ε, μπορούμε να τα εξετάσουμε σε μια έναν απλό κατακαιρματισμό συμφερόντων στην Ευρώπη ω προ τη γεωγραφική του έκθεση. Αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ πιο περίπλοκα τα πράγματα από αυτό. Τα ζητήματα στην Ανατολή δεν αφορούν μόνο την Πολωνία και τα κράτη τη Βαλτική. Στο Νότο, επίση, τα προβλήματα δεν αφορούν μόνο την Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα ή την Τουρκία. Υπήρξε μια πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση από, την, ε, από το Ίδρυμα Pew Research και έχουμε εξετάσει εν συντομία αυτά τα αποτελέσματα και στη ΣΥΠΑ έγινε δημοσκόπηση, αλλά και στην Ευρώπη. Ζήτησαν λοιπόν από το ευρύ κοινό πόσο τους απασχολεί, πόσο τους προβληματίζουν ορισμένες ε, προκλήσεις άμυνας και ασφάλειας. Και στην Πολωνία, για παράδειγμα, κάτι το οποίο μας εξέπληξε ιδιαίτερως, θεωρούσαμε ότι θα υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη ε, ιεράρχηση προτεραιοτήτων ως προς τις προκλήσεις. Όντως, το 71% των Πολωνών πολιτών θεωρούν ότι η Ρωσία είναι πολύ σημαντική απειλή, το 73% θεωρούν ότι ο ISIS είναι πολύ σημαντική απειλή για την Πολωνία. Επομένως, ως προς την αντίληψη, ως προς την πολιτική, το στρατηγικό σχεδιασμό, βλέπουμε ότι είναι ευρύτερα τα πράγματα. Και η Τουρκία έχει τη δική της έκθεση, είναι ιδιαίτερη περίπτωση. Και μέχρι πρόσφατα νομίζω ότι εξέτασαν περισσότερο το θέμα της Ρωσίας ε, και όχι τα υπόλοιπα. Θεωρούσαν ότι θα αλλάξει η προοπτική τους, αλλά αν σκεφτείτε τη Μαύρη Θάλασσα, την Ανατολική Μεσόγειο, εδώ έχουμε περιοχές που ουσιαστικά και η Ανατολή και ο Νότος μας απασχολούν. Νομίζω ότι θα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και δεν θα επιληθεί μάλλον στην οδοκορυφή, ούτω ώστε οποιασδήποτε έχουμε για την άμεση απόκριση από το ΝΑΤΟ εν γέννη συνδέονται με όλα αυτά και αφορούν και πολύ και τον Νότο και για την Ιταλία και για τα υπόλοιπα μέλη νομίζω. Τρίτο και τελευταίο στοιχείο. Πίσω από αυτό το προσκήνιο έχουμε και κάποια άλλα ευρύτερα ζητήματα. Πολλά από αυτά αφορούν τις ΗΠΑ. Μία από τις ευκαιρίες που θα προκύψουν από τη Σύνοδο είναι μια ευκαιρία και δυνατότητα για τον πρόεδρο Ομπάμα και για άλλους υψηλούς αξιωματούχους τον ε, ΗΠΑ να μιλήσουν με κάθε έμφαση ε, για την σημασία των ε, ιδανικών αυτών σχέσεων για την άμυνα και την ασφάλεια. Είναι μια πολύ σημαντική συζήτηση αυτή στις Ηνωμένε Πολιτείε για τον επιμερισμό των βαρών, για την ε, συμμετοχή μας ε, στην Ευρώπη, όλα αυτά τα σημαντικά ζητήματα. Πριν ανησυχούσαμε για το πώς οι Αμερικανοί στρέφονται προς την Ασία. Τώρα είναι πολύ ευρύτερο το ζήτημα. Τώρα λέμε Πώ ουσιαστικά με το έτος των εκλογών στο οποίο θα περάσουμε θα μπούμε σε μια αποσύνδεση από την Ευρώπη. Δεν ξέρω πώ θα γίνει, αλλά έχουμε το φαινόμενο Τραμπ από αυτή την άποψη και θα πρέπει να το εξετάσουμε και πολύ σοβαρά. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν για να καταδείξουμε ότι είναι σημαντικός φορέας το ΝΑΤΟ ε, και ότι διασκεδάζει σημαντικές ανησυχίες του κοινού θα είναι κάτι θετικό. Για τις ΗΠΑ αυτό είναι ωφέλιμο σε πολλά επίπεδα. Υπήρξε μία επαναστατική αλλαγή σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή ε, αμυντική συνεργασία. Στο παρελθόν υπήρξε μεγάλος ε, σκεπτικισμός, αλλά τώρα βλέπουμε ότι οι μεγαλύτεροι υπερασπιστές ε, της ευρωπαϊκής στρατηγικής συνεργασίας, αμυντικής συνεργασίας, είναι οι Αμερικανοί. άλλα πράγματα που βλέπουμε ότι είναι πραγματικά θετικές εξελίξεις, ότι το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν πάλι πολύ πιο σοβαρά το θέμα της συνεργασίας. Αυτό το βλέπετε και στο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Παγκόσμια Στρατηγική που μιλάει και κάνει σημαντικό λόγο για το ΝΑΤΟ, κάτι το οποίο μας προκαλεί έκπληξη. Και τέλο, κάτι το οποίο αποτελεί πρόκληση και για το ΝΑΤΟ και για την Ευρωπαϊκή Ένωση ω προ ζητήματα αρμοδιότητα αλλά και δημοσίου ενδιαφέροντο, υπάρχει συζήτηση κατά πόσο η τρομοκρατία είναι υπαρξιακό κίνδυνο. Ενδεχομένω όχι πρακτικά, αλλά πολιτικά. Εάν οι συμμαχίε δεν αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα, θα τεθούν πολύ σημαντικά και δύσκολα ερωτήματα και στους πολιτικούς. Αν δείτε, λοιπόν, αν κοιτάξουμε προς το μέλλον, μετά τη Βαρσοβία, θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην καταπολέμηση της δημοκρατίας. Θα μείνω εδώ, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Thank you, sir. Ευχαριστούμε. Και τώρα, να ξεκινήσει η συζήτηση. Ο κύριος Στετίνα. κύριε Πρόεδρε, Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε για τις αναλύσεις σας και τους τρεις ομιλητές. Ειδικά τώρα που αναφύονται νέοι κίνδυνοι για την ασφάλεια. Είναι πολύ σημαντικό να μιλήσουμε για τη συνεργασία μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και με μεγάλη χαρά βλέπω ότι και οι τρεις να το αναφέρετε. Βλέπω και οι τρεις να το αναφέρετε. Λοιπόν, Προς τον κύριο Τζέιμι Σέι, μία ερώτηση. Μιλήσατε για τον υπηρετικό πόλεμο και ότι στη Βαρσοβία θα γίνει λόγος, θα συζητήσετε με την κυρία Μογκερίνη για τους υπηρετικούς πολέμους και τις διαδικασίες και τις στρατηγικές που θα πρέπει να αναπτυχθούν για να αντιμετωπιστεί ο υπηρετικός πόλεμος. κατά τύχη χθε κάναμε εδώ μία ακρόαση με τον κύριο Πόρτμαν, που είναι επικεφαλής της, του τμήματος Stratcom, που δημιούργησε η κυρία Μογκερίνη. Τον ρωτήσαμε διάφορα πράγματα για την χρηματοδότηση που υπάρχει στη διάθεσή μας και τι εργαλείες έχει το τμήμα αυτό στη διάθεσή του. Και είδαμε ότι υπάρχουν τεράστιες διαφορές. Η Ρωσία, Φερρυπίν, ξοδεύει εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια κάθε μήνα για υβριδικό εξοπλισμό. Η Stratcom εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προσωπικό 9 δεκάτομα μόνο. Ο υβριδικός πόλεμος είναι πολύ επικίνδυνος. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ε, Ρωσία. Και τις στάσεις αυτές που έχει. Βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι σε θέση να αμυνθεί αποτελεσματικά. Το ΝΑΤΟ είναι σε καλύτερη θέση για να υπρασπιστεί τα συμφέροντά μα σε περίπτωση που υπάρξει υβριδικό πόλεμο. Και κάτι άλλο, ε, κύριε Σέι. Μιλήσατε για τις περικοπές στον αμυντικό προϋπολογισμό ε, και την ανικανότητά μας να τηρήσουμε τις ε, δεσμεύσεις που είχαμε λάβει για τις δαπάνες. Και η τσεχική δημοκρατία δεν είναι σε θέση να σεβαστεί αυτή τη δέσμευση που είχε αναλάβει για το 2% των αμυντικών δαπανών. Επομένω, λοιπόν, θέλω να σα κάνω εξή ερώτηση για αυτό το θέμα. Πιστεύετε ότι οι σημερινέ προκλήσει που αντιμετωπίσουμε είναι τόσε, ούτω ώστε να πρέπει να αυξήσουμε τον, τις αμυντικές μας δαπάνες. Νομίζω, εγώ προσωπικά, ότι οι προκλήσεις είναι τόσο γνωστές. Και αν αυτές οι προκλήσεις δεν μας δίνουν τις, την απαραίτητη αιτιολογία για να αυξήσουμε τις αμυντικές, ε, να αυξήσουμε τις αμυντικές μας τότε τι θα μας το δώσει. Ο Τζέφαν Βανόρντεν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα ήθελα να πω καταρχά ότι με μεγάλη χαρά σας καλούμε εδώ και είμαι μεγάλος οπαδός του German Marshall Fund. Είδαμε και τον κύριο Πόρκα μαζί μας, ο οποίος συμμετείχε στη σημερινή μας στο Λονδίνο και πάντα μεγάλη μου χαρά να βλέπω τον Τζέμι Σέιν πραγματικά ε, εδώ και χρόνια τον γνωρίζουμε και τον βλέπουμε σε διάφορες περιστάσεις να είμαστε σαφείς ότι η, ο επόμενος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής ε, τον είπα, θα επιμείνει οι Ευρωπαίοι να συμβάλλουν πιο πολύ στην άμυνα το θέμα της κατανομής των παρών. Προσεκτικά θα έλεγα ότι ας μην υποθέσουμε ότι αυτό θα σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δημιουργήσει αυτό το σκέλος της αμυντικής ικανότητας που λείπει και ότι θα ήταν αξιόπιστος εταίρος ε, τον είπα. Νομίζω ότι το αντίθετο ενδεχομένω να συμβεί. Θα είναι μάλλον ε, αφηρημένο αυτό, αφηρημένη αυτή ως οργάνωση και ο κύριος Πούτιν πολύ θα χαρεί να δει τη διαμορφώση δύο πόλων στην Αντιατλαντική Συμμαχία. Το μήνυμα λοιπόν που θα ήθελα να στείλω στους φίλους μας από την άλλη πλευρά ε, του Ατλαντικού είναι ας μην προκληθεί σύγχυση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ευρωπαίων Συμμάχων. Και γι' αυτό χαίρομαι ιδιαίτερως ε, που στο ΝΑΤΟ δεν φανταζόμαστε ότι η απάντηση στα προβλήματα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά αυτή την γελία υπόθεση της ε, Συνεργασία Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Μα τα ίδια έθνη συμπεριλαμβάνονται και τώρα χρειάζονται μακροσκελείς μηχανισμοί για να μιλάνε για τα ίδια πράγματα, τα ίδια έθνη μεταξύ του, Είναι πραγματικά γελίο αυτό. Και εγώ θα είμαι ο πρώτο, ο οποίο ε, θα αναγνωρίσει ότι υπάρχουν πολλοί τομεί στους οποίου δεν θα πρέπει να δραστηριοποιείται ο ΝΑΤΟ σε ό,τι αφορά τα ήπια μέσα, σε ό,τι αφορά ε, το θέμα της διαχείρισης πολιτικών κρίσεων και υπάρχουν πάρα πολλά σημεία όπου θα μπορούσε να είναι χρήσιμη η Ευρωπαϊκή Ένωση με στοχευμένου πόρου, να είναι πιο αποτελεσματική. Θα πρέπει να επικεντρωθεί στα πράγματα λοιπόν αυτά, παρά να παίζει άλλα παιχνίδια. Φρίκη μου προκαλεί το γεγονός ότι το ΝΑΤΟ ε, εμπλέκεται σε τέτοια ευρωπαϊκά, μάλλον σε τέτοια προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μεσόγειο. Μου θυμίζει αυτό τη διαδικασία ε, και όσα έγιναν ε, στη δεκαετία του 90 που είχαμε δύο στόλους να ε, πηγαίνουν πάνω κάτω στη Μεσόγειο, στην Ευρετική του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά μέχρι ότου αποφασίστηκε το λογικό, το μοναδικό λογικό πράγμα να αναλάβει το ΝΑΤΟ τις δραστηριότητες αυτές. Άρα θεωρώ και αυτό που με ανησυχεί σε ό,τι αφορά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ είναι ότι το ΝΑΤΟ ασφαλώς παίζει το παιχνίδι αυτό, γιατί οι εκπρόσωποι του ΝΑΤΟ, οι πρωθυπουργοί οι οποίοι παραβρίσκονται, είναι οι ίδιοι οι οποίοι συμμετέχουν και σε άλλα φόρα και προασπίζονται όλα αυτά τα στοιχεία υπέρ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Προφανώ λοιπόν χρησιμοποιούν και την ίδια γλώσσα όταν βρίσκονται σε σύνοδο του ΝΑΤΟ, να μην το ξεχνάμε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, γνωρίζετε ποια είναι η απόψή μου το θέμα αυτό. Το πιο προβληματικό στοιχείο του Brexit ίσως να προκαλέσει έκπληξη δεν είναι το αποτέλεσμα και η έκβαση η οποία ήταν η πλέον ευκταία θεωρούσα. Δεν ήθελα να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μία από τις μεγαλύτερες παρενέργειες είναι ότι το Ηνωμένο Βασίλειο σε δύο-τρία χρόνια δεν θα είναι πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως αποτρεπτικός και παράγοντας ε, συγκράτησης και θα επικρατήσουν οι πιο αυτονομιστικές γερμανικές, αν θέλετε, ε, τοποθετήσεις. Αυτή θα είναι λοιπόν η μεγαλύτερη ανησυχία μου. Και δύο-τρεις μικρές ερωτήσεις έχω να θέσω. Αναφέραμε την Τουρκία ήρθε στο εμπαρόδο. Η Τουρκία αποτελεί μια τεράστια ανησυχία. Ανησυχία θα έλεγα, γιατί είναι βασικός σύμμαχος κλειδί του ΝΑΤΟ και είδαμε την φρικτή αυτή και αποτρόπαια α, τρομοκρατική επίθεση στην Τουρκία, στο, στην Κωνσταντινούπολη. Έχουμε και τα σύνορα με την ε, Συρία. Πρόκειται για μια χώρα που έχει τεράστια εσωτερικά προβλήματα. Ποια είναι λοιπόν η άποψή σας για την ενίσχυση της συμμαχίας με την Τουρκία. Πώς μπορούμε παραπάνω να δεσμεύσουμε στους κόλπους της Ιδρυτικής Συμμαχίας και την Τουρκία για να είμαστε βέβαιοι ότι θα συνεχίσει να αποτελεί αξιοπιστό και σταθερό εταίρο. Και κατά δεύτερον, αυτό που λείπει νομίζω από τις συζητήσεις μας είναι το ότι το ΝΑΤΟ θα πρέπει να εξηγήσει καλύτερα στο ευρύ κοινό το γιατί θα πρέπει να επενδύσουμε στην άμυνα και γιατί έχουμε ενέπλε δυνάμει. Γιατί πιστεύω ότι υπάρχει μια ολόκληρη γενιά νέων ανθρώπων που απλά δεν το καταλαβαίνουν. Το μόνο που βλέπουν είναι ότι οι ένοπλε δυνάμει δημιουργούν προβλήματα στον κόσμο και δεν καταλαβαίνουν γιατί πραγματικά χρειαζόμαστε να αντιμετωπίσουμε τι προκλήσει και του κινδύνου. Ένα πιο συγκεκριμένο θέμα προ εσένα, Τζέιμι. Μιλήσαμε για την αξιοπιστία τη συμμαχία. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι τα μηνύματα, τα σήματα τα οποία στέλνουμε σε ανθρώπους όπως ο Πούτιν. Και αυτοί δεν κοιτάνε μόνο τα προφανή και τα επιφανειακά, αλλά αυτό που κρύβεται και πίσω από τις κάποιες ενέργειες. Ένα λοιπόν στοιχείο είναι η ενδυνάμωση, η, μεγαλύτερη α, επένδυση σε α, δυνατότητες, σε ικανότητες της συμμαχίας. Και τέλος, θα υπάρξει κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα, κάποια συγκεκριμένη έκφαση ως αποτέλεσμα της Συνόδου. Είπατε τα διάφορα για την επίδειξη α, κοινού χαρακτήρα και ενότητας, αλλά θα υπάρξει κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα προκειμένου ο κόσμος να καταλάβει ότι μάλιστα μιλάμε σοβαρά. Ευχαριστώ η κυρία Νικολάη, λέει η πρόεδρος. Ευχαριστώ. μερικούς, εδώ και μερικούς μήνε, μάλλον όλοι εξετάζουμε αυτό το πολύ σημαντικό και διάσημο ζήτημα της κατάρριψης του ε, ρωσικού αεροσκάφους από την Τουρκία. Όμως θα είναι δύσκολο να εξετάζουμε και να δούμε πώς η Τουρκία, η Ρωσία, το Ισραήλ θα, κάνουν μια, θα συνάψουν μια τέτοια συμμαχία. Δεν ε, γνωρίζουμε πολλά για το τι σημαίνει αυτή η συμμαχία. Θα είναι μόνο για την καταπολέμηση του ISIS, είναι μια στρατηγική συμμαχία για τη Μαύρη Θάλασσα, γιατί βλέπουμε μια αλλαγή ε, σε ό,τι αφορά τη Ρωσία, αλλά δεν είναι πραγματική αλλαγή για μένα, γιατί ε, συνεχώς ε, ασχολούνται με τη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο, γιατί χρειάζονται τις δύο περιοχές. Ε, έχω ακούσει πολλούς ε, αξιωματούχους να κάνουν λόγο για την ε, σύμβαση του Μοντρέ. Μετά βλέπω την αντίδραση της Βουλγαρίας στη ρουμανική πρόταση να έχουμε μία μόνιμη δύναμη στη Μαύρη Θάλασσα. Η δική σας γνώμη ποια είναι για αυτή την κατάσταση. Το δεύτερο ερώτημά μου. ως προς ε, τις ευρωπαϊκές δυνάμεις, την ευρωπαϊκή ικανότητα. Ακόμα και για το ποιος θα είναι μετά ο, ο νέος Αμερικανός πρόεδρος, ο Τραμπ ή η κυρία Κλίντον. Όπως και να έχει, το θέμα της ευρωπαϊκής ε, στήριξης και συμμετοχής ε, θα τεθεί επιτάπητος και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Δυστυχώς, χάσαμε σημαντική ικανότητα, τη Βρετανική. ποιες είναι οι σκέψεις σας ό,τι αφορά τις μελλοντικέ φιλοδοξίες ε, της Ευρώπης ε, στο πλαίσιο της ε, πολιτικής ασφαλείας. Και το τρίτο ερώτημά μου αφορά τον Κάφκασο και πιο συγκεκριμένα τη Γεωργία. Δεν βλέπουμε ξεκάθαρα ποια είναι η κατάσταση της Γεωργίας. Ποια είναι η γνώμη σας σε ό,τι αφορά την κατάσταση σε αυτή τη χώρα, ε, η οποία συμμετέχει περισσότερο από τις χώρες της περιφέρειας. Ευχαριστώ κύριε Βαλέρο. Ευχαριστώ πολύ. Έχω ένα ερώτημα για τον ε, Γενικό Γραμματέα για τον στόχο του 2% του ΑΕΠ. Γιατί το θέμα δεν είναι μόνο οικονομικό. Δεν είναι μόνο πόσα χρήματα δίνει, αλλά και τι αποτελέσματα έχει για αυτά τα χρήματα. Και δεν υπάρχει καμία χώρα που πραγματικά να έφτασε το στόχο ω προ τα αποτελέσματα. Τι θα κάνετε λοιπόν για να αλλάξετε αυτή την ισορροπία. Εγώ προέρχομαι από μια χώρα που δεν είναι μέλο του ΝΑΤΟ και δεν έχουμε το στόχο αυτό του 2% του ΑΕΠ για την άμυνα. Όμως, Εντάξει, τώρα έχουμε μια νέα κατάσταση ε, ως προς την ασφάλεια. Πήραν περισσότερα χρήματα, αλλά το Κοινοβούλιο είναι αυτό που αποφασίζει τι πόροι θα δοθούν σε κάθε τομέα πολιτικής. Και όταν το Κοινοβούλιο αποφασίσει ότι τώρα αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε περισσότερα για την αμάνη, άμυνα, συγγνώμη, ε, αυξάνουμε τις αμυντικές μας δαπάνες. Αλλά το 2% δεν σημαίνει τίποτα στην ουσία για την ικανότητα που τελικά θα αναπτύξει κάθε χώρα. Τι θα κάνετε λοιπόν για να αλλάξετε αυτή την κατάσταση, γιατί δεν είναι το παν τα χρήματα. Με τα χαίρομαι που λέτε ότι τώρα πράγματι μάθατε το μάθημά σας από την Λιβύη και το Ιράκ, ότι πάντα θα πρέπει να υπάρχει μια επιπλέον στρατηγική. Όταν κλείνει μια αποστολή, μια επιχείρηση πρέπει να δούμε τι θα γίνει μετά. Δεν το αφήνουμε έτσι στην τύχη και ελπίζουμε τα πράγματα να πάνε καλά. Από ό,τι βλέπω λοιπόν ε, μάθετε το μαθημά σας και στο μέλλον ε, θα σκέφτεστε ε, και λίγο πιο προοπτικά. Ένα άλλο ερώτημα τώρα, σε ό,τι αφορά τον ΝΑΤΟ και τον Frontex. Νομίζω ότι είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση όταν αρχίζουμε να αναμειγνύουμε στρατό και μεταναστευτικό. Δεν είναι στρατητικό αυτό το πρόβλημα. Ε, με τα χαράς ε, να βοηθήσετε τον Frontex για να σώσετε ανθρώπινες ζωές, αλλά αυτό θα πρέπει να είναι το βασικό σημείο εστίασης. Ενώ τελικά βλέπουμε στην πράξη ότι θέλουμε τους μετανάστες να μην έρχονται εδώ. Αυτό είναι το κύριο ζήτημα για τον Frontex και παρεμπιπτόντως να σώσουμε και ανθρώπινες ζωές. Εντάξει, κανένα πρόβλημα αν θέλετε να βοηθήσετε να σωθούν ανθρώπινες ζωές, αλλά δεν πρέπει να στρατιωτικοποιήσουμε το μεταναστευτικό υπερβολικά. Ευχαριστώ. Κύριε Τζιούρεκ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Όταν ε, μιλούμε για την Ευρώπη, όχι για τη Μεσυνατολή, εξετάζουμε πώς θα ενισχύσουμε τις ε, αμυντικές μας δυνατότητες σε περίπτωση επίθεσης από τη Ρωσία. Βλέπουμε τι έχει συμβεί τα τελευταία 20 χρόνια. Δεν είχαμε συγκρούσεις με συμμάχους ε, του ΝΑΤΟ. Πρέπει να εξετάσουμε τι συμβαίνει στα πιο ευάλωτα μέλη μας, ε, τις χώρες της Αλλά τα τελευταία 20 χρόνια είδαμε ε, μία παρέμβαση στη, στην εσωτερική πολιτική σκηνή περισσότερο και από την Τσετσενία και από τη Βοσνία και από την Ουκρανία. Πρόκειται για περιοδικές ε, συγκρούσεις ε, που εξυπηρετούν εξωτερικά συμφέροντα. για να μεγιστοποιήσουν τη μεγαλύτερη στρατηγική του 20ου αιώνα, την κατάρρευση της Βιωτικής Ένωσης. Καταστροφή, συγγνώμη, του 20ου αιώνα. Επομένως, αν δούμε τι συνέβη τα τελευταία 20 χρόνια, πρέπει να είμαστε έτοιμοι και για νέες προκλήσεις. Και να δούμε πώς θα διασφαλίσουμε αυτή την ισορροπία και τη σταθερότητα στις σχέσεις μας. Όταν προκύπτουν αυτές οι νέες συγκρούσεις, μπορούν να λάβουν διαφορετικό χαρακτήρα, δεν είναι όλες στρατητικές. Είδαμε ότι η Ρωσία ε, ουσιαστικά καταδίκασε την ε, ε, οικονομική προσέγγιση της Αρμενίας προς τη Δύση. Υπάρχουν δηλαδή πολλοί τρόποι να το κάνει αυτό η Ρωσία. Τώρα δύο ερωτήματα για την Ουκρανία. Πού καταλήγουμε, ποιο είναι το συμπέρασμά μας ως προς την προσάρτηση της Κρυμαίας. Για 5, 10, 15 χρόνια στο μέλλον Ε, θα λέμε ότι δεν μπορούμε να αποδεχθούμε την προσάρτηση της Κρυμαίας. Δεν υπάρχει επιλογή. Πρέπει να το επαναλαμβάνουμε συνεχώς. Όμως, η προσάρτηση της Κρυμαίας σημαίνει μεγαλύτερη σταθερότητα για τη Ρωσία στην περιφέρεια. Η Ρωσία ήθελε να βελτιώσει, να ενισχύσει τη θέση της στην ευρύτερη περιφέρεια και τώρα έχουμε μια ειδική κατάσταση στη Γεωργία. Γιατί οι σύμμαχοί μας εκεί φυλακίζονται. Όμως η κοινωνία είναι ιδιαίτερα φιλοευρωπαϊκή, φιλοδυτική μάλλον. Έχουμε διαφόρους ε, αναλυτές, όπως ο Τζορτ Φρήμαν, που λένε ότι η στήριξή μας προς τη γεωργία είναι μόνο θεωρητική επιχάρτου και ότι η Ρωσία θα αυξήσει την επιρροή της εκεί. Επομένω, τίθεται το ζήτημα. Έχουμε την πρόθεση να υπερασπιστούμε τη γεωργία. Γιατί μετά την Κρυμαία, τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Όμω, όταν υπήρξε εισβολή στη Γεωργία, θα μπορούσαμε να αντιδράσουμε. Είχαμε μία φιλικά διακείμενη ε, κυβέρνηση στη Γεωργία που δέχτηκε επίθεση, μία ξεκάθαρα φιλοδυτική ε, κυβέρνηση. Πρέπει να απαντήσουμε λοιπόν σε αυτά τα ερωτήματα, να εξετάσουμε και να προβλέψουμε νέε συγκρούσει σε τομεί και περιοχέ που θα επιλέξει ο, ο Πούτιν. Όχι περιοχέ που εμεί απαραίτητα είμαστε έτοιμοι και προετοιμασμένοι να υπερασπιστούμε. Αυτό είναι κέριο ζήτημα. Και δεύτερον, στο ευρωπαϊκό προσκήνιο, αν θέλετε, την περιοχή του Καλίνιγκραντ. Εμείς έχουμε έναν ε, άλλο όρο στην Πολωνία για αυτή την περιφέρεια. Το θέμα είναι ο ρόλος όμως αυτής της περιοχής που είναι ιδιαίτερα στρατιωτικοποιημένη. Εμείς θέλουμε να επιστρέψουμε στις ε, φυσιολογικές ε, σχέσεις διαλόγου με τη Ρωσία. Όμως δεν θα πρέπει να κάνουμε λόγο για αυτή την ε, κατάσταση στο Καλίνιγκρατ που δεν είναι φυσιολογική. Έχουμε λοιπόν μια τέτοια περιοχή, ένα θύλακα αν θέλετε, που απειλεί την Πολωνία και τα κράτη της Βαλτικής και το καθεστώς της και ο στρατικός της χαρακτήρας και ρόλος θα πρέπει να μας απασχολήσει. Αυτά είναι παραδείγματα μεγαλύτερου στρατηγικού βάρους. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να δούμε πώς ε, θα βελτιώσουμε την άμυνα και ασφάλειά μας και πώς θα αποδυναμώσουμε τους αντιπάλους μας. Θα ήθελα να ακούσω κάτι και για τα σχόλια Φρίντμαν. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχουν άλλα σχόλια. Από ό,τι βλέπω. Θα ήθελα και εγώ λοιπόν με τη σειρά μου να θέσω ένα ερώτημα στους καλεσμένους μας. Όχι πρόεδρο, ως πρόεδρος, αλλά ως απλή ευρωβουλευτής μέλος αυτής της ε, υποεπιτροπής. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη που άκουσα να αναφέρεται η μελέτη που προετοιμάστηκε από ένα κέντρο. Στην ε, μελέτη αυτή υπάρχουν διάφορες, διάφοροι πίνακες που δείχνουν ότι η θέληση των λαών της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυτή που ξέρουμε. Έχουμε μία σύγκριση μάλιστα ανάμεσα στη στάση Ευρωπαίων και Αμερικανών και ανάμεσα στο πώς οι δύο διαφορετικές κοινωνίες, δηλαδή η ευρωπαϊκή και η αμερικανική, είναι έτοιμοι να χρηματοδοτήσουν την οικοδόμηση στρατιωτικού δυναμικού. Τι κάνουμε εμείς στην Ευρώπη και τι κάνουν οι Αμερικανοί. Και νομίζω ότι οι πολιτικές αποφάσεις που θα λάβουμε εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη ενοποίηση στην αμυντική πολιτική και μεγαλύτερες, μεγαλύτερη συνεργασία και πιο στενή συνεργασία με τον ΝΑΤΟ. Σε περίπτωση που γίνει το Brexit, που βγει τελικά η Βρετανία, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι πολλά κονδύλια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διοικητικού σκοπούς, παρά για την οικοδόμηση της ειρήνης. Υπάρχουν κάποιες διοικητικές λειτουργίες που αλληλεπικαλύπτονται, ας πούμε. Να μην πάμε χρήματα εκεί. Εσείς τι άποψη έχετε, στρατηγέ. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ η διπλωματική γλώσσα, εμένα πρέπει να σας πω. Και νομίζω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούμε μια φρασιολογία η οποία δεν αυξάνει, δεν κλιμακώνει την ένταση. Εδώ μιλούσαμε για περιορισμό της Ρωσίας. Και περιορισμό των αυτοκρατορικών της βλέψεων. Η αναχέτηση των αυτοκρατορικών της ε, βλέψεων. Διερωτώ με, είμαστε αξιόπιστοι. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι η Ρωσία θα κάνει αυτή τις μικρές έντασεις, ε, θα κάνει αυτές τις μικρές, ε, μικρές επιθέσεις αυτή, αυτής χαμηλής έντασης πόλεμου, ε, που δεν ξέρω είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε τη συμπεριφορά της Ρωσίας ε, αποτελεσματικά. Ας ξεκινήσουμε τώρα με, τους, ε, με τις απαντήσεις των καλεσμένων μας, ο στρατηγός ΣΥΑ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χίλια ευχαριστώ. Πολλές ερωτήσεις. Ε, και εμείς το ίδιο κάνουμε όταν έρχονται διάφοροι να μας ενημερώσουν τους λέμε κάντε ερωτήσεις, λέμε στα μέλη μας κάντε ερωτήσεις, αλλά ε, μην υπερβείτε τα δύο λεφτά. Ε, εδώ πέρα βλέπω υπάρχει μια μεγαλύτερη ανεκτικότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, εν πάση περιπτώσει, εγώ θα χρησιμοποιήσω περισσότερο χρόνο βέβαια, αλλά μην με κατηγορήσετε μετά ότι αποφεύγω ερωτήσει. Τέλο πάντων, θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι μπορώ καλύτερο. Καταρχά, για την ειρήνη. Ε, Βεβαίω, η Ρωσία έχει επενδύσει πάρα πολύ καλά στα κρατικά μέσα ενημέρωση Ε, το ΝΑΤΟ και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, ξέρετε ότι έχουμε, εδώ πληρώνουμε ας πούμε ανθρώπους ε, για να είναι επιθετικοί μόνο στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. και φυσικά μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και άλλη όψη του νομίσματος που, υπάρχει, που είναι ότι δεν υπάρχει καν αλήθεια. Μην προσπαθείτε να πιστέψετε τίποτα γιατί μπερδεύουμε τόσο πολύ τα, τα πράγματα, ε, με τόσο πολλές ιδέες κτλ. Ε, ε, και η Ρωσία μάλιστα μας, ε, ακριβώς αυτό λέει. Κοιτάξτε, διαδίδουμε τόσες ε, ας πούμε ειδήσει και τα λοιπά που δεν πρέπει να πιστεύετε τίποτα και ούτε αυτά που σας λένε κυβερνήσει σας βέβαια. Κοιτάξτε, όχι, υπάρχουν ε, κάποια στοιχεία. Εμείς πρέπει να σπάσουμε τους μύθους. Θα πρέπει να φανούν ξεκάθαρα ε, τα στοιχεία. Ε, πέρυσι, θα θυμάστε, ότι οι Ρώσοι έλεγαν δεν έχουμε επιχειρήσεις ε, και δυνάμεις στην ε, Ουκρανία. Είναι μύθος. Εμείς όμως ε, εμφανίσαμε τις δορυφορικές εικόνες και δείξαμε τις δυνάμεις τους με τα αρχικά τους, με τα τάγκ τους και αποδείξαμε ότι υπάρχουν. Και μας βοήθησαν όλες οι κυβερνητικές οργανώσεις, το Ηνωμένο Βασίλειο, που κάνουν ε, γεωεντοπισμό, ε, που κάνουν έρευνα στα μέσα, τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης και δικτύωσης κτλ. Ε, για να αποκαλύψουν την αλήθεια. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι, είναι να ρίχνουμε, ας πούμε, μία χιονοστιβάδα, ας πούμε, νέων. Ε, υπόθηκε από Αμερικανό πρόεδρο Ντρούμαν ότι μπορεί να ξεγελάσεις λίγους ε, για μεγάλο χρονικό διάστημα ή πολλούς για μικρό χρονικό διάστημα. Δεν μπορεί να γελά τους πάντες για πάντα. Έτσι. Προσοχή όμως, ε, τα ΜΜΕ, ε, τα μα μας πεθαίνουν γιατί υπάρχουν περικοπές, υπάρχουν τόσες περικοπές και πιέσεις στον προϋπολογισμό διώχνονται δημοσιογράφοι. Αν θέλετε πλουραλιστικά ε, ΜΜΕ, που είναι το τελευταίο χειρό ενάντια στην προπαγάνδα, πρέπει να κοιτάξετε τι μπορούμε να κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να προστατεύσουμε ουσιαστικά του δημοσιογράφου, τα ΜΜΕ, από τι μαζικέ εμπορικέ πιέσει που υφιστάμεθα. Φυσικά ε, έχουμε τι οργανώσει μα, ε, θα πρέπει να κοιτάξουμε πώ μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τα κοινωνικά μέσα, μην το ξεχνάτε. Η δική μου γενιά πιστεύει ότι πρέπει να κοιτάμε την ε, συνέντευξη τύπου, α πούμε, στο CNN, τότε που εγώ ήμουν εκπρόσωπο του ΝΑΤΟ. Έτσι, αυτό αρκούσε, α πούμε. Αλλά όχι, τώρα θα πρέπει να αποκεντρώσουμε λιγάκι. Θα, πρέπει να δούμε πώ μπορούμε να ενισχύσουμε του ε, ανθρώπου μα, ούτω ώστε να περάσουν την δική μα άποψη ε, στα ΜΜΕ. Ε, μπορεί, αν συνεχίσουμε, ας πούμε, ένα άτομο να μιλάει και να εκπροσωπεί την ε, οργάνωση, δεν μπορεί να είναι το άτομο αυτό παντού. Δεν μπορεί να κλωνοποιηθεί, ας πούμε. Κάτι θα χάσουμε, κά, κάποιον θα ξεχάσουμε. Ε, Επομένω, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε του πόρου μα καλύτερα. Αλλά η αίσθησή μου είναι ότι αυτό το είδου η προπαγάνδα μπορεί να είναι και αντιπαραγωγική τελικά για τη Ρωσία ε, επίση η προπαγάνδα ε, γίνεται όλο και λιγότερο πιστευτή όσο περισσότερο συνεχίζεται, καθώς ο κόσμος αναγνωρίζει πραγματικά τι θέλει να διαδώσει. Θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι για το τι κάνουμε εμείς για να ε, παρεμποδίσουμε το μονοπόλιο των ΜΜΕ και τι μπορούμε να κάνουμε ε, ε καλό είναι, ας πούμε, ε, να τιμωρούνται όσοι λένε ψέματα. Ε, ε, πρέπει να έχουμε επιτροπέ για να εξετάσουμε παράπονα. Σε, αυτά τα, σε αυτά τις επιτροπές δεν θα πρέπει απλώς να απλώς να λέμε ας πούμε ε, τα νέα ας πούμε σαν να είμαστε μηχανήματα κτλ. Να σπάμε τους μύθους θα πρέπει. Θα πρέπει να επαληθεύουμε ας πούμε τα στοιχεία ειδικά ε, τις πιο εξωφρενικές ας πούμε διατυπώσεις αυτές που να τις πάμε. Δεν είναι το θέμα να κάνουμε προπαγάνδα στην προπαγάνδα των άλλων. Είναι τι μπορούμε να κάνουμε ούτως ώστε να διατηρήσουμε ε, ποιοτικά και πλουραλιστικά ε, ΜΜΕ στις ε, κοινωνίες μας. Ο Τζέφρι έκανε πάρα πολλές ε, πολύ σημαντικές ερωτήσεις. Έξι, τρομερές ερωτήσεις, ε, πολύτιμες. Ξέρεις τη θέση μου για πολλά. για τον Brexit καταρχάς. Ε, οποιοδήποτε και είναι το αποτέλεσμα, ό,τι άποψη και αν έχουμε, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κρατήσουμε το Ηνωμένο Βασίλειο εμπλεκόμενο στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Το θέλουμε, νομίζω. Το Ηνωμένο Βασίλειο είπε ξεκάθαρα ότι σε ό,τι αφορά τη συνοκορφή του ΝΑΤΟ ε, είναι αξιόπιστο ε, σύμμαχο που θα τηρήσει όλε τι δεσμεύσει και έχει αναλάβει μεγάλε δεσμεύσει. Είναι μεγάλο παίχτη ε, σε αυτό το σχέδιο ετοιμότητα. ανέφερα τα αεροσκάφη, ε, τη διοίκηση, τη μεραρχία κτλ. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει το 50% της ευρωπαϊκής, των ευρωπαϊκών αμυντικών δαπανών. Θα ήταν μεγάλη απώλεια αν το χάναμε, ας πούμε, αυτό. Ε, και εδώ, ας πούμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάθε λόγο να κάνει ό,τι μπορεί ε, για να πείσει το Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί η Ευρωπαϊκή Αμυντική Συνεργασία χωρίς το Ηνωμένο Βασίλειο, ας τα πούμε τα πράγματα έξω από τα δόντια, ε, το Ηνωμένο Βασίλειο ε, έχει και πολλές πληροφορίες, υπηρεσίες πληροφοριών, έχει ε, ένα στρατιωτικό δυναμικό που ελάχιστες ευρωπαϊκές χώρες έχουν αυτή τη στιγμή. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ΚΠΑ, ε, στο, στο παρελθόν, ας πούμε, εμπλέξαμε την Νορβηγία, τον Καναδά, την Τουρκία, νομίζω. Ε, κοιτάξτε όμως ε, την α, συμβολή των Βρετανών στις α, στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μεσόγειο, ας πούμε, στις ε, ναυτικές επιχειρήσεις, συγγνώμη, στη Μεσόγειο έχει ένα πλοίο εκεί πέρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχει κάθε λόγο να τίνει χείρα προ το Ηνωμένο Βασίλειο. Και κάτι πολύ σύντομο, Τζέφρι. Νομίζω ότι η συνεργασία Ευρωπαϊκή Ένωση ΝΑΤΟ είναι ακόμη πιο σημαντική αν θέλουμε να κρατήσουμε το Ηνωμένο Βασίλειο ε, στο ΝΑΤΟ. Ε, θα πρέπει να είναι πιο μέσα στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Και είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει καλή σχέση με το ΝΑΤΟ, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα χτίσουμε μια γέφυρα με το Ηνωμένο Βασίλειο. Ενώ στο παρελθόν ξέρει ότι το ΝΑΤΟ μιλούσε πάντα για τη συνεργασία Ευρωπαϊκή Ένωση και η κυρία Μογκερίνη είναι πολύ καλή, ε, ε, σε αυτό, ήταν πολύ καλή σε αυτό το έγγραφο Παγκόσμια στρατηγικής. Ε, στο μέλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάθε λόγο να τίνει χείρα προς τον ΝΑΤΟ, τόσο ώστε να διατηρήσει την εμπλοκή του Ηνωμένου Βασιλείου. Επίση, ε, αμυντική συνεργασία Ευρωπαϊκή Ένωση ΝΑΤΟ. Ε, καλό είναι να συνεργαστεί και, και να μην κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίω αυτά που έχει κάνει το ΝΑΤΟ. Και δεν έχουμε ατελείωτο χρήμα και αυτό που ξοδεύουμε το ξοδεύουμε συνετά. Νομίζω ότι για μένα η αρχή είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ θα πρέπει να συνεργαστούν στο Νότο, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να αφήσει την αμυντική, τη συλλογική άμυνα α, στα ανατολικά, ας πούμε, ε, στην αποκλειστική ε, ας πούμε, αρμοδιότητα του ΝΑΤΟ, έτσι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει τι μπορεί να, ε, τι μπορεί να κάνει για τα ανατολικά. Υπάρχει η θαλάσσια διάσταση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κάνει πολλά. Ε, με την ε, με την αστυνομία και την ε, ε, χωροφυλακή. Γιατί ε, ο μικρό πόλεμο, σημαίνει, ο πόλεμο χαμηλή ένταση, σημαίνει ότι ελέγχει τα σύνορά σου. Ούτω ώστε να μην διεισδύουν διάφοροι, α πούμε, από τα σύνορα. Μπορούμε να δείξουμε και φαντασία. Πρέπει να δούμε να κάνουμε, και να κάνουμε πράγματα ρεαλιστικά. Το ΝΑΤΟ, α πούμε, Φερρυπίν, έχει ξεκινάει να προσφέρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ομάδε μάχη. Ε, Ας δούμε λοιπόν ε, αυτές τις ευκαιρίες που έχουμε. Μου κάνω μια άλλη μια ερώτηση για την Τουρκία και την Κεντρική Μεσόγειο επίσης. Α, τι μπορεί να κάνει το ΝΑΤΟ για να βοηθήσει. Χρειαζόμαστε να έχουμε διπλούς στόλου, Όχι, Τζέφρι. Αλλά μπορούμε να βοηθήσουμε, ας πούμε, με, ε, με, με τη διοίκηση που ε, προσφέρουμε κτλ. Ε, Τζέφρι, η, με, η Μεσόγειος θα έχει το πρόβλημα αυτό για τα πολλά επόμενα χρόνια. Ε, το ΟΗΕ θεωρεί ότι ο πληθυσμός της Ασίας θα διπλασιαστεί ε, μέχρι το 2050. Ξέρουμε ότι η οικονομική μετανάστευση σπρώχνει και πιέζει και θα είναι εκεί ε, πολύ μετά την, το καταλάγιασμα ας πούμε, του προσφυγικού κύματος. Και πρέπει να ελέγξουμε τη Μεσόγειο που είναι τεράστια περιοχή. Έχουμε την Ανατολική Μεσόγειο, ας πούμε. Βλέπετε πώς τα, οι προσφυγικές ροές μπορούν να αλλάξουν, ας πούμε, και να ακολουθήσουν άλλους δρόμους. Ε, Τουρκία. Τι θα βοηθούσε. Ε, η Τουρκία ε, καταλαβαίνει τώρα νομίζω πια ότι το ISIS ε, την απειλεί και την ίδια, όχι μόνο εμάς, το αποδεικνύει τίνοντας χείρα προς το Ισραήλ. Το, η Τουρκία χρειάζεται την προστασία του ΝΑΤΟ. Το απέδειξε η ανάπτυξη που κάνουμε στα πλαίσια του Patriot. Για το θέμα της Κύπρου, επίσης καλό θα ήταν να βοηθήσουμε γιατί θα βοηθήσει και τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ ποιοι θα είναι οι επιχείροι τίτλοι από την Βαρσοβία. Θα, ε, θα ανακοινώσουμε την ανάπτυξη τεσσάρων νέων ε, ταγμάτων ε, και τη δίκησή τους. Θα ανακοινώσουμε την, το φυσικό δυναμικό ε, των, της αντιπυραυλικής άμυνας. Ε, ένα μεγάλο ε, κομμάτι του ΝΑΤΟ στο Νότο θα προστατεύεται. Επίσης θα έχουμε τη νέα θέση για τη Γερτική Μεσόγειο με, την, με τις επιχειρήσεις Endeavor. Έχουμε τη δήλωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δήλωση ναι, αλλά πολιτικά είναι πολύ σημαντική. Θα ανακοινώσουμε τον εξυγχρονισμό του στόλου μας το 2035 με, όλη αυτή αυτό το νέο δυναμικό θα ανακοινώσουμε μια στρατηγική για να αντιμετωπίσουμε με του, τους μη κρατικού ε, φορεί που έχουν όπλα μαζική καταστροφή ε, ε, στο, Νότο. Θα καλωσορίσουμε το Μαυροβούνιο, θα του δείξουμε ανοιχτή πόρτα. Ναι, το ανακοινωθέν σίγουρα θα έχει μάλλον 120 παραγράφους. οι πιο ενδιαφερόμενοι μπορούν να διαβάσουν όλα αυτά, ας πούμε. Αλλιώς επιλέξετε. Λοιπόν, και για να σταματήσω, το 2%. Έχετε δίκιο. Το θέμα δεν είναι το, να, το θα ξοδεύει, το, σε τι θα είναι. Ε, τα μισά μέλη του ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή ε, στρέφονται προς μία αύξηση ε, αμυντικών δαπανών ε, και δεν θα ξοδεύουν όλο το ποσό αυτό σε αυτά που θέλουν αυτοί μόνο, αλλά και στι προτεραιότητε του ΝΑΤΟ. Θέλουμε πιο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για να βοηθήσουμε αυτού να κάνουν και σωστέ επιλογέ, τα μέλη μα δηλαδή. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορεί πάντα να λε και το κάνουν αυτό κάποιοι σύμμαχοί μα τα τελευταία χρόνια. Α, δεν χρειάζεται να ξοδεύουμε παραπάνω. Γιατί θα αναδιοργανωθούμε και θα ξοδεύουμε τα ίδια, αλλά πιο σοφά. Σωστό αυτό, καλό. Αλλά αυτό έγινε και μία δικαιολογία για να μην ξοδεύει κανεί παραπάνω. Και δεν πήραμε, δεν αυξήσαμε έτσι το δυναμικό μα με αυτόν τον τρόπο. Τελικά, όπω τα περισσότερα στη ζωή, αν θέλει το προϊόν, θα πρέπει να κάνει και την επένδυση και να βάζει το χέρι στην τσέπη. Να πολιτείε εξοδεύουν πολύ περισσότερα, πολύ πάνω από το 2% και θα είναι πολύ δύσκολο να κρατήσουμε, ας πούμε, ε, μια καλή ε, διατλαντική σχέση εάν εμείς ξοδεύουμε συνέχεια το 73% και καλύπτουμε το 73% του προπολογισμού του ΝΑΤΟ. Ε, ίσως λοιπόν το 2% είναι μια χονδροειδή, ας πούμε προσέγγιση, αλλά πολιτικά είναι σημαντικό ότι αυτό, και να πούμε ότι αυτό που χρειάζεται για να ε, αναπτυχθούμε. Η εμπειρογνώμη μας μας λέει ότι αν όλοι ε, ξοδεύουμε αυτό το 2% θα φτάσουμε στο να μπορούμε να σε δυναμικο ανεφοδιασμο ανεφοδιασμού αέρος-αέρος όλα τα αμυντικά στοιχεία και εξοπλισμό που χρειαζόμαστε για την άμυνά μα. Και αυτό θα ήταν επωφελέ για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, δεν θα ήταν μόνο επωφελέ για τον, για τον ΝΑΤΟ. Ε, με βάση του υπολογισμού μου, απάντησα μόνο το 1 τρίτο των ερωτήσεων και αφήνω του συναδέλφου για να απαντήσουν στα υπόλοιπα 2 2-3 τρίτα. Ευχαριστώ. Θα Σα ευχαριστούμε κύριε Γενική Γραμματέα. Δυστυχώ, ναι, είναι πραγματικά συναρπαστική αυτή η συζήτηση, αλλά δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάρκεια μα. Να δώσουμε το λόγο στον ε, στρατηγό Πόλκο. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Η συζήτηση ήταν ε, για θέματα τα οποία έχουμε συζητήσει επί μακρόν. Για την αναχέτηση της Ρωσίας θα ήθελα να απαντήσω. Η Ρωσία ασφαλώς ε, ε, διαρκώς εκμεταλλεύεται τις αδυναμίες του συστήματος μας. Ε, η Ουκρανία αρχικά μετά τα, οι πράσινοι στρατιώτες στην Ουκρανία με όλα τα ψέματα που συνοδεύουν αυτή τη διαδικασία και αυτά προφανώς πάνε χέρι-χέρι με την προπαγάνδα των δραστηριότητες. Αυτός ο πόλεμος λοιπόν μέσω της προπαγάνδας αρχικά δεν έγινε αντιληπτό απαραίτητα από τη Δύση. Πρόκειται για προκλήσει. Προκλήσει οι οποίε είναι οριακέ λοιπόν σήμερα. Αν λοιπόν η αντίδρασή μα ενώπιον τέτοιων προκλήσεων διαμορφώνεται με τον τρόπο τον εξή, ότι επιβεβαιώνουμε ότι η Ρωσία αποτελεί εταίρο και όχι απειλή και ότι ο Πούτιν αποτελεί τμήμα του της λύσης. Όλα αυτά προφανώς οδηγούν σε κλιμάκωση της, των προκλήσεων από πλευράς της Ρωσίας. Το σημαντικό είναι να εξαγάγουμε και τα μαθήματα από τα παθήματα του παρελθόντος. Τι έκανε ο Ρίγκαν σε ό,τι αφορά τις προκλήσεις αυτές. Αυτά οδήγησαν στην κατάρρευση της Ευρωπαϊκής ε, της Ένωσης τελικά. Και μας απασχολεί και η ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στο Καλίνιγκραντ. Και αυτό αποτελεί στρατιωτική πρόκληση. Και ε, το θέμα δεν είναι μόνο ε, μία πλήρη στρατιωτική σύγκρουση. Δεν θέλουμε μόνο αυτό να προσωμιώσουμε, αλλά θέλουμε να προσωμιώσουμε και απειλές ή πουλές οι οποίες μπορεί να προελθούν από τα ανατελικά σύνορα και τις οποίες επίσης θα πρέπει να μπορούμε να επιλύσουμε. Η Ρωσία στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ λοιπόν ε, ενδεχομένως ε, να πει ότι πρέπει από κοινού να αντιδράσουμε και μάλιστα δυναμικά. Και αυτό που θα ήταν πάρα πολύ ε, επικίνδυνο θα ήταν να καταρρεύσουν και στο ιστορικό τους οι δομές μας. Γιατί για την ανάπτυξη ευρωπαϊκών δυνάμεων θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο, μάλλον αν γίνει αυτό με τρόπο που ε, θα διασπάσει την ενότητα των δυνάμεών μας, αυτό θα το εκμεταλλευτεί ε, ο Πούτιν και προφανώς θα εκδηλώσει έτσι περαιτέρω την κατάστασή μας. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό. Όχι μόνο, μάλλον σίγουρα να ε, ανταπεξέλθουν στις, να ανταποκριθούν στις ευθύνες τους τα μέλη του ΝΑΤΟ και όπου υπάρχουν ε, ε, ελλείψεις να καλυφθούν τα προβλήματα. Και στο σημείο αυτό θα ήταν απαραίτητη και η διεξαγωγή ενό ελέγχου, όπω έγινε στη Γερμανία, για να εντοπιστούν καταρχά οι ελλείψει αυτέ και μετά να γίνει α, η κάλυψη των κενών αυτών. Φυσικά χρειάζονται και ασκήσει, στι οποίε ε, κάθε χώρα θα πρέπει να αποστέλει επαρκεί δυνάμει, επαρκεί στρατιώτε, προκειμένου πραγματικά να υπάρχει ενότητα και ομόνια στο ιστορικό της, του ΝΑΤΟ, γιατί οι κίνδυνοι είναι προφανείς, ξέρετε, δεν είναι δυνατόν να μένουμε σε επίπεδο ασφών ικανοτήτων, οι οποίες δεν είναι σε καμία περίπτωση συγκεκριμένε Και σε ό,τι αφορά τι χρηματικέ ε, επενδύσεις, θα πρέπει να υπάρξει συγκεκριμένη απόδοση των πόρων. Ή Ιταλία δεν θα πετύχουμε τίποτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Γιάννη Λέσνερ. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι τα περισσότερα έχουν ήδη σχολιαστεί, όμως ε, να δείξω κάποια ακόμα. Για το θέμα των αμυντικών δαπανών, θεωρώ ότι όποιο και αν ε, κερδίσει τι εκλογέ ε, στι ΗΠΑ, δεν θεωρώ ότι έχει και πολλέ πιθανότητε ο Τραμπ, αλλά όπω και να έχει. Αυτή η έννοια τη ε, άσκηση ψηλών πιέσεων προ την Ευρώπη για τον επιμερισμό των βαρών και των δαπανών δεν θα φύγει. Είναι ένα μακρόχρονο ζήτημα δεν θα επιληθεί. Μπορεί όμως να πάρει μια νέα τροπή. Δεν το συζητήσαμε, αλλά καθώς θα επανεξετάσουμε το θέμα της πυρηνικής στρατηγικής, το οποίο είναι μια πολύ σημαντική πτυχή της σύνδεσής μας με τον ΝΑΤΟ, κατευθείαν ερχόμαστε στο ζήτημα των ε, συμβατικών, ε, στρατιωτικών και αμυντικών ικανοτήτων. Εμείς αυτό θέλουμε, να ε, επαναλάβουμε τη δέσμευσή μας ακριβώς για αυτή την ικανότητα. Τίποτα δεν θα μας χαροποιήσει περισσότερο στις ΗΠΑ. Δεν θα φύγει λοιπόν αυτό. Για την Τουρκία πολλά έχουν ήδη υποθεί. Η Τουρκία μπορούμε νομίζω και ελπίζω να πούμε ότι είναι η μοναδική χώρα αυτή τη στιγμή στο ΝΑΤΟ που κάποιο ε, του πυροβολεί στα σύνορα. Που δέχεται δηλαδή καθημερινά τέτοιε επιθέσει. Και αν δείτε τα, τα σχέδια ετοιμότητα τα οποία θα πρέπει να έχει το ΝΑΤΟ και τα προβλήματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσει τα επόμενα χρόνια, τα περισσότερα αφορούν τα τουρκικά σύνορα ή κάπως με κάποιον τρόπο εμπλέκουν την Τουρκία. Είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστούμε είτε το πρόβλημα στην Ανατολή, ιδίω στη διάσταση τη Μαύρη Θάλασσας, είτε στο Νότο, χωρί στενή συνεργασία ασφάλεια με την Τουρκία στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Οι Τούρκοι βεβαίως έχουν και αυτοί δουλειά να κάνουν προς αυτό, γιατί την τελευταία δεκαετία περίπου η Τουρκία δεν νομίζω ότι τα είχε όλα αυτά στο επίκεντρο του στρατηγικού της σχεδιασμού. Όμως καθώς αναπτύσσονται και επιδεινώνονται αυτά τα προβλήματα, ε, προσπαθούν να βελτιώσουν τις σχέσεις τους με τη Ρωσία, το Ισραήλ, γι' αυτό θα θέλουν να έχουν και αυτή τη διασφάλιση με τον ΝΑΤΟ. Αλλά ποτέ δεν υπήρξε και ποτέ δεν θα είναι μια ε, εύκολη σχέση έτσι κι αλλιώς, όπως και με εκείνη την αεροπορική βάση. Τέλος, για τη μείωση του κινδύνου, νομίζω ότι είναι ε, ένα κρίσιμη σημασία καθήκον μετά τη Βαρσοβία σε ό,τι φορά την μείωση του κινδύνου. Βλέπουμε ότι οι πιθανότητες ε, ατυχημάτων, τυχαίων δηλαδή περιστατικών, ιδίω στη Μαύρη Θάλασσα, στη Μεσόγειο κτλ αφορά μια αυτή τη μείωση κινδύνου από τακτικής άποψης, αλλά και για το πώς θα ανοίξουμε και πάλι αυτό τον χαμένο διάλογο για το τι εννοούμε με σταθεροποίηση και αποσταθεροποίηση. Και αυτό ενδεχομένως είναι πιο αμερικανικό ζήτημα και συζήτηση μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, όπως ήταν στον ψυχρό, πόλεμο, αλλά δεν το έχουμε κάνει εδώ και πολύ καιρό και θα ήταν προς όφελος όλων να ξεκινήσει και πάλι αυτή η συζήτηση. Σας ευχαριστώ και για αυτό το τελευταίο σχόλιο σας. Το θεωρώ εξαιρετικά ενδιαφέρον και αρκετά καινούριο και καινοτόμο. Σας ευχαριστώ. Κυρίε και κύριοι, έτσι φτάνουμε στο τέλος της σημερινή ε, συζήτησης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, διακεκριμένους μας ε, ομιλητές. Σας ευχαριστώ πολύ. Η επόμενη συνεδρία θα λάβει χώρα στις 13 Ιουλίου, μετά την ε, Σύνοδο της Βαρσοβίας. Ελπίζουμε λοιπόν να έχουμε και νεότερα τότε. Σας ευχαριστώ.